Liebe Kolleginnen und Kollegen, συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε γιατί στην κοινή μας ε, συνεδρίαση έχουμε μόνο έναν περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε μια άλλη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και της δικής μας ε, προκειμένου να εξετάσουμε τα δύο σχέδια έκθεσης όσον αφορά το Europass και το θέμα της νέας στρατηγικής της ε, δεξιότητες για την Ευρώπη. Λοιπόν, ε, υπάρχει μόνο ένα σημείο της ημέρησης διάταξης, έγκριση των πρακτικών. Έχετε παρατηρήσεις? Εάν όχι, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, ανακοινώσεις της Προέδρου. Σήμερα το πρωί έχουμε μετάφραση στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, σουηδικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, λιθουανικά, πολωνικά, σλοβακικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Επίσης θα ήθελα να σε επισημάνω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται από το διαδίκτυο και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από το, φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Πουατιέ κατόπιν πρόσκληση της κυρίας Μωρίν Σατιέ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα τμήμα της συνεδρίασής μας. Γιατί είναι νέοι οι οποίοι ε, μελλοντικά, σε λίγο μάλλον, θα πρέπει να μπουν στην αγορά εργασία. Άρα είναι θέματα που του αφορούν. Και ελπίζω η συζήτηση αυτή να κινήσει το ενδιαφέρον σας και ενδεχομένως να πάρετε και κάποια ρεθίσματα. Εν πάση περιπτώσει καλωσορίσατε στις επιτροπές μας. Äh, Πριν ε, μπούμε στις δύο εκθέσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα διαδικαστικά θέματα. Για τη δεύτερη έκθεση ε, υπήρξε παράκληση για την ε, μετάθεση της προθεσμίας υποβολή, της ημερομηνίας υποβολής καταθέσεων τροπολογιών. Εξετάσαμε το θέμα και είδαμε ότι το πολύ μπορούμε να βάλουμε μέχρι τις 6 Απριλίου στις 12 ε, το μεσημέρι. Ε, στην, ε, για την έκθεση Europass οι ημερομηνίε μένουν όσα έχουν, έτσι όπως έχουν προταθεί. Δηλαδή, εδώ είναι 30 Μαρτίου, 12 η ώρα και η εξέταση των τροπολογιών στις 25 Απριλίου. Το γεγονό ότι εδώ πρόκειται για μια ε, νομοθετική, έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, σχετίζεται με τον ορισμό της ημερομηνία για, ε, για την εξέταση των τροπολογιών και άρα λοιπόν δεν μπορεί να αναβληθεί περαιτέρω, αλλά για, το, για τη δεύτερη έκθεση Skills Agenda θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να δώσω τη συνάδελφο Μαρίτα Ούσκοφ ως ε, συμπρόεδρο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι καλό είναι να αρχίσουμε δίνοντας το λόγο στους εισηγητές απευθείας για το θέμα αυτό. Στον κύριο Μάν, λοιπόν, θα δώσω το λόγο από την Επιτροπή Απασχόλησης και μετά τον κύριο Μαλινόφ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που έχουμε δύο καλές επιτροπές, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα πετύχουν κοινά αποτελέσματα. Όσον αφορά τους, εμάς τους δύο εισηγητές, η συνεργασία μας ήταν πολύ επικοδομητική. Βλέπετε εδώ το καρπό της προσπάθειας. Ε, καταθέσαμε 25 κοινέ τροπολογίες και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τόσο καλή συνεργασία μεταξύ δύο επιτροπών ε, ούτω ώστε να μπορεί να χαραχθεί ενδεχομένω μια κοινή πολιτική γραμμή. Εν πάση περιπτώσει και δύο προσανατολισόμεθα προς μια συνένεση. Ε, η υποστήριξη του Europass είναι διαφυσβήτητη. Ε, έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο και η ιδέα θα πρέπει να εξεγχρονιστεί και να βελτιωθεί. Μας βρίσκει σύμφωνος. Θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο όπου η, όσοι αναζητούν εργασία αλλά και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ε, αλλά αν 15 χώρες έχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν, ε, αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε ως εξή. Είναι υπερβολικά γρήγορος ο ρυθμός της διαδικασίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί εστιάζονται οι επιφυλάξεις ε, γιατί αυτό το οποίο μέχρι στιγμή έχει επιτευχθεί στις, στο επίπεδο των δεν θα πρέπει να υπονομευθεί. Θέλουμε να διατηρηθεί η πολυφωνία ε, και ένα Europass έχει νόημα μόνο εφόσον δεν υπερφορτωθεί με όρους και προϋποθέσεις, αλλά είναι εύχριστο. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια βήματα, τους να το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε, ένα, έχουμε εθνικά κέντρα Europass ήδη από το 2004 και εκεί ε, ε, ε, διατυπώνονται οι δεξιότητες στο επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει και η ΕΣΚΟ στην Κομισιόν. Τι είναι αυτό το σύστημα. Μια, ένα σύστημα ταξινόμησης για τις δεξιότητες και τις ειδικότητε. Γιατί αυτή η κοινή βάση θα πρέπει να προσαρμοστεί σε όλο το φάσμα των των χωρών μελών. Πρόκειται για ένα project το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί στο επίπεδο των χωρών μελών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε... Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει εδώ. Ένα άλλο σημαντικό σημείο. Έχουμε ε, υπηρεσίες συντονισμού, εθνικές ομάδες εμπειρογνώμων του Europass που εργάζονται πολύ αποτελεσματικά, που πραγματικά εργάζονται με επιτυχία. Δεν είναι ένας μηχανισμός ε, παρακόλλησης, ε, αλλά ε, είναι μια προσπάθεια να μετατραπεί η Ευρώπη σε ένα εργαστήριο εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Και εδώ εντάσσεται και το Europass. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε πραγματικά να ανοίξει ένα διάλογο με αυτές τις υπηρεσίες. Τέλος, χρειαζόμαστε μια λύση προς μια πλούστευση αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά τι ημερομηνίε, ε, έχω κάποιε επιφυλάξει. Χθε το βράδυ, στι διαπραγματεύσει και στι συζητήσει με το Συμβούλιο, έμαθα ότι από το Συμβούλιο θα γίνει μια προσπάθεια επεξεργασία στι 6 Απριλίου και θα ήταν ε, ανόητο αν δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί η παρούσα εργασία του Συμβουλίου, γιατί αλλιώς θα δυσκολέψουν διαπραγματεύσεις ε, σε τριμερές επίπεδο. Άρα λοιπόν να μην διατηρήσουμε τις 30 Μαρτίου γιατί στις 6 Απριλίου θα έχουμε νέα αποτελέσματα. Ίσως θα μπορούσαν να δουν οι συντονιστές ε, πώς μπορεί να αναβληθεί παρόλα αυτά ε, η ημερομηνία μέχρι τις 10 Απριλίου. Μπορούν, πιστεύω, να το κάνουν οι συντονιστές και οι βοηθοί μας. Ε, τουλάχιστον να πάμε μέχρι τη 10η Απριλίου για να είναι επικαιροποιημένο το ντοσιέ και να γίνουν σωστά οι διαπραγματεύσεις. Ε, χαίρομαι με προκαταρτικά για την συζήτηση με τον συνάδελφο Μαλινόφ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαλίνοφ, έχετε το λόγο από την Επιτροπή Πολιτισμού. Αν ο κύριος Μάν έχει δίκιο, αν πράγματι συνεργαστούμε, δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω και ειδικότερα αν υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις, πρέπει οπωσδήποτε να τις ε, αντιμετωπίσουμε, να τις απομακρύνουμε. Θα ήθελα να εξηγήσω ποια ακριβώς είναι το πρόβλημα για τους συναδελφούς. Έχουμε το αρχικό πλαίσιο του Europass που είναι ένα σύνολο εγγράφων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να γίνει μία πλατφόρμα παροχής υπηρεσίας με κάποιες αλλαγές και παράλληλα υπάρχει και συνένεση ότι το παλιό πλαίσιο είναι ε, επαρκές. Οπότε ε, πώς μπορεί κάτι που είναι πολύ επιτυχημένο να το αλλάξει κανείς ε, σε κάτι ακόμη πιο, πιο, πιο επιτυχημένο, κάνοντας μάλιστα αλλαγές που μπορεί να ε, μη βελτιώσουν την κατάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, τους ε, συμβούλους μας και τους ε, βοηθούς μας, γιατί με την ταπεινή μου εμπειρία πρέπει να πω ότι αυτή η διατύπωση ξεκίνησε με πάρα πολύ έντονη αλλά πολύ ε, καλά αιτιολογημένη αντίσταση από τα κράτη-μέλη. Ο αριθμός ήταν πολύ υψηλότερος από την, αρχηγή, από την αρχική, ε, από την δυνατότητα που υπήρχε για την κίτρινη κάρατα. Όμως στη συνέχεια ε, είπαν ακριβώς τι ήθελαν. Υπήρξε μια γενική συνένεση ότι η αναθεώρηση χρειάζεται και ήταν αρκετά ειλικρινοί τα κράτη-μέλη να πούν, στο να πούν ακριβώς τι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ποιες είναι οι ανησυχίες τους. Η υποχρεωτική χρήση της ΕΣΚΟ αυτό είναι κάτι καλό αλλά όχι πλήρως ανεπτυγμένο και ίσως ε, στο μέλλον, αν είναι επιτυχές, θα έπρεπε να αναπτυχθεί περαιτέρω και ήταν σαφές ότι το θέμα της διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για αυτά, ότι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σήμαινε πολύ ε, περισσότερους κινδύνους, οικονομικούς κλπ. Οπότε ο τίτλος εργασίας ήταν η αναθεώρηση του Europass. Ε, πράγματι, κάναμε την αναθεώρηση, αλλά ε, τότε νόμιζα ότι είχαμε μια καλή βάση ε, διαπραγμάτευσης. Όμως όσοι ήθελαν πιο φιλόδοξο ε, πιο φιλόδοξη αλλαγή. Ε, είναι λίγο δυσαρεστημένοι. όμως τα κράτη-μέλη που και αυτά είχαν, κάπως, είχαν εκφράσει κάποιες ανησυχίες έχουν καταφέρει τελικά να αποδεχθούν το συμβιβασμό. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν με όλα αυτά τα οποία μας έχουν προταθεί, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο και αν η ΕΣΚΟ ήταν επιτυχής, ε, υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες, οι τεχνολογικές αλλαγές ε, ελπίζουμε ότι δεν θα μας υποχρεώσουν να κάνουμε τίποτε πολύ νωρίτερα. Πάντως η κατάσταση τώρα είναι καλή μετά από μια πολύ δύσκολη διαδικασία ε, ε, διατύπωσης. Πιστεύω ότι η αναθεώρηση του Europass είναι επιτυχής. Αυτό που θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής είναι ότι για τους ε, σπουδαστές που είναι εδώ είναι μια τυπική διαδικασία μιας ε, πολύ φιλόδοξης και κάπως ρηψοκίνδυνης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε πολύ καλά αιτιολογημένες απόψεις από τα κράτη-μέλη και βρήκαμε έναν συμβιβασμό που ήταν τελικά ο μοναδικός δυνατός τρόπος ε, η αποφυγή των συγκρούσεων, η αποφυγή των κινδύνων και πίσω από τις ιδέες ε, και τα λόγια ε, των ε, εθνικών ε, κέντρων δεξιοτήτων ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο και μερικές φορές όχι τόσο χρήσιμο να υπάρχει απόλυτη εναρμόνιση. Θα πρότεινα να, προχω... να συστήσω διαδικαστικά στο τέλος. Ε, νομίζω τώρα θα πρέπει να διευκρινίσουμε το περιεχόμενο. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις των δύο επιτροπών και θα ξεκινήσω με τη συνάδελφο Μαρίτα Όσκουκ για δύο τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγητές. Είναι σαφές ότι αντιμετωπίσατε τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας και γενικά μπορώ να πω ότι συμβαδίζουμε Νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την σύνδεση με την πρωτοβουλία ΕΣΚΟ που βρίσκεται σε ε, προπαρασκευαστικό στάδιο και δεν ξέρουμε αυτός, αυτή η διασύνδεση πώς θα ισχύσει έμπρακτα. Νομίζω ότι το Europass θα πρέπει να είναι ένα εθελούσιο μέσο διαφάνειας και να βελτιώσουμε αυτό που ήδη είναι να μην μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή το Europass και να αντιγράψει τα προϋπάρχοντα. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει αυτά τα ε, εθνικά συστήματα συντονισμού έτσι ώστε να υπάρχουν ε, μεταδεδομένα για το συντονισμό των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να δούμε ε, όμως ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες, γι' αυτό θα υποβάλουμε και τροπολογίες. Ε, υπάρχουν θέμα που, θέματα που ως προς το Europass ότι δεν είναι φιλικό προς το χρήστη και ότι δεν φτάνει τους, στους κύριους ε, χρήστες του, ενδυνάμει χρήστες. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Θα πρέπει να δούμε και τη διατύπωση σε σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους ε, εταίρους και, τους, ε, και αυτούς όλους όσους συμπλέουν με το σχέδιο. Είναι ένα καλό σημείο κίνησης. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μόνικα Σμέρκοβα για την, ε, από την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Κατά την τελευταία μας ε, συνεδρίαση, στο τέλος, είπα ότι χρειάζεται μία βαθύτερη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τη σωστή νομοθεσία χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία των ε, πληροφοριών. Δεν νομίζω ότι έγινε αυτή η ανάλυση εις βάθος όπως θα έπρεπε, που είναι ύψης της σημασίας. Γι' αυτό η πρόταση της είναι πολύ φιλόδοξη, υπερβολικά φιλόδοξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί υπάρχουν τάχιστες αλλαγές στην αγορά εργασίας και στις νέες τεχνολογίες. Ε, αν δούμε πώς λειτουργεί το Europass στα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι κανένας δεν ξέρει για την ύπαρξή του. Θα πρέπει να ε, γίνει γνωστό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια, στις, στους οργανισμούς ε, παροχής επαγγελματικών συμβουλών και ούτω καθεξής. Οι συνάδελφοί μου έχουν μία σειρά τροπολογιών που σχετίζονται με τα εξής. Η πρόταση της Επιτροπής δεν λέει σε ποιον απευθύνεται το Europass. Επίσης θα πρέπει να μιλάμε για κοινωνικούς εταίρους και οργανισμούς νεολαίας, να μην μιλάμε για εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων είναι αυτό που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι το ΕΣΚΟ σε σχέση με τις δεξιότητες ιδιαίτερα, διότι αυτό το πλαίσιο δεν έχει οριμάσει. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε το ε, ρόλο της άτυπης ε, μάθησης μαζί με άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως αυτό το πυρήνα αλληλεγγύης. Νομίζω ότι δεν είναι ένα ευέλικτο μέσο το ΕΣΚΟ. Τώρα, σε σχέση με τις δεξιότητες και τις ικανότητες, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουμε έναν ορισμό των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων πριν προβούμε σε αυτή την ταξινόμηση, διότι δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων μας δίνει έναν ορισμό. Επειδή δεν θέλω να είμαι επικριτικός, θα ήθελα να πω ότι το έγγραφο της ε, Επιτροπής είναι ενδιαφέρον γιατί θέλει να αναβαθμίσει το Europass, το οποίο άρχισε να ισχύει από το 2004. Ελπίζω με τις τροπολογίες μας να κάνουμε πιο θελκτικό το πλαίσιο, το οποίο είναι ένα χρήσιμο μέσο σε αυτό το τομέα των ε, ικανοτήτων και προσόντων. Δελεαστικό μέσο όμως δεν σημαίνει ότι θα προβάλλουμε μία πλημμυρίδα προς τις ε, εθνικές αρχές μέσα στα πλαίσια του γραφειοκρατικού φόρτου. Το Europass θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο μέσο παροχής πληροφοριών σε σχέση με τις ε, δεξιότητες και τα επαγγέλματα. Θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που χτυπάω με το σφυρί, αλλά πραγματικά υπάρχει περιορισμός χρόνου και θα πρέπει να τηρούμε τα περιθώρια ομιλίας για να μην πιεστούμε υπερβολικά. Η Γιάννα Τσιτεύσκα από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εκ μέρου του συναδέλφου από την Επιτροπή Πολιτισμού. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα δικά του λόγια. Αγαπητοί τι εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα περιορίσω τα σχόλιά μου στο σχέδιο έκθεσης που ο εισηγητής μας παρουσιάζει σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που διαπιστώνω ότι φαίνεται ότι είναι κοινέ οι ανησυχίες και προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν με επικοδημητικές τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Η ECR υποστηρίζει τροπολογίες που αφορούν το σεβασμό της ε, ε, αρχής της κούσιας ε, οικοδόμησης της Ευρώπης. Μέσω των τροπολογιών θέλαμε να κάνουμε κούσια τη χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου ειδικοτήτων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών μέσω του Europass και τη διαγραφή του άρθρου 6 του πλαισίου, γιατί δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ταξινομήσεις ως βάση για το Europass εφόσον δεν έχει αναπτυχθεί πλήρω ούτε έχει εγκριθεί από τι χώρε μέλη. Τέλο, οι τροπολογίε που αφορούν το ζήτημα του κόστου και τη σχέση με την αποτελεσματικότητα θα υποστηριχθούν από την ECR. Ε, η κυρία εργάστηκε σκληρά για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ε, και γι' αυτό οι τροπολογίε από την Επιτροπή Πολιτισμού θα είναι περιορισμένε. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Όπως σας είπα, χαιρετίζω την προσπάθεια αναθεώρησης της Ευρώπης γιατί είναι αναγκαίο να εξυγχρονιστεί αυτό το εργαλείο και θέλουμε να πετύχουμε το τομείς οι οποίες, ε, ε, ότι υπάρχουν τοπίες που θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτισμού. Θα πρέπει να ε, είναι θελούσια συμμετοχή. σημαντικό είναι η πλατφόρμα αυτή να είναι προσβάσιμη από άνθρωπα με αναπηρία τα οποία δυσκολεύονται ε, πολύ περισσότερο ε, και χρειάζονται μια υποστήριξη προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και υπό την έννοια αυτή θα θέσω εγώ τις δικές μου, θα υποβάλω τις δικές μου τροπολογίες. Τώρα θα έρθουμε στην ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής, ε, θα έρθουμε στην ε, εκπρόσωπο από το ΑΛΔΑ, από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Διάβασα την έκθεσή σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για την εξαιρετική έκθεση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε σημεία. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στη σχέση κόστους-οφελίας, να βρούμε μία καλή εξισορρόπηση ε, ως προς το διοικητικό και χρηματοδοτικό ε, φόρτο με βάση τη σχέση αυτή ε, κόστους-οφελίας. Το Europass θα πρέπει να είναι ένα θελούσιο μέσο για όσους αποζητούν εργασία και για τους εργοδότες που το επιθυμούν δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από αυτούς που το επιθυμούν. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία που βοηθά τους νέους, ιδιαίτερα όταν δεν ξέρουν πώς να γράψουν ένα βιογραφικό, βιογραφικό ή να ορίσουν τα προσόντα τους. Δεν θα πρέπει να είναι το έσκο υποχρεωτικό, γιατί αυτή τη στιγμή η Επιτροπή προβαίνει στη σύστασή του. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή ε, διαβούλευση και μία διακυβερνητική βάση ανάπτυξης του Europass για τους τελικούς χρήστες. Θα πρέπει όμως να έχουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων έτσι ώστε αυτές οι υπηρεσίες να είναι υψηλής ποιότητας και να δούμε κατά πόσο χρειάζονται και ποιες αλλαγές χρειάζονται σε σχέση με την κατάρτιση θεωρώ ότι χρειάζεται καλύτερη διατύπωση με βάση τις εθνικές πρακτικές. Θα υποβάλω ορισμένες τροπολογίες, αλλά θα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι το... η έκθεση αυτή είναι σχεδόν τέλεια. Και δεν το λέω συχνά αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χουντής έχει τώρα το λόγο από την ΚΟΕ και την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ τους συνεισηγητές. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον και τις παρουσιάσεις τους. Σημείωσα τα θέματα που υπάρχουν διαδικαστικά και άλλα. Θα ήθελα όμως να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι για το Europass και την αναβαθμισμένη πλατφόρμα θα μπορούσε να πει κανείς αρχικά ότι δεν διαφωνεί αν είναι ένα εργαλείο που θα ωφελούσε και θα διευκόλυνε τους εργαζόμενους, τους νέους που μας παρακολουθούν τώρα, στην αναζήτηση εργασίας με βάση τα προσόντα τους και θα τους εξασφάλιζε αξιοπρεπείς και ποιοτικέ θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Επίσης, θέλω να σας θυμίσω ότι εκεί που εμφανίζεται ότι είναι ένα ουδέτερο, ένα τεχνοκρατικό, θα έλεγε κανείς, εργαλείο, ότι δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία, αλλά τα εργαλεία αυτά ε, εφαρμόζονται για να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις. Κατά τη γνώμη μου αυτό το ρόλο θέλει να παίξει και επιτελεί το Europass και πολύ περισσότερο η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του Europass που μάλλον μονοπολεί τη συζήτησή μας σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας, κατά την άποψή μας, <clears throat> αυτή η τεχνική, αυτή η διαδικασία, αυτό το εργαλείο καλείται να υποστηρίξει τεχνικά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Το κέντρο βάρους μεταφέρεται στην αγορά εργασίας και στην πολιτική δεξιοτήτων. Για τις δεξιότητες θα τα πούμε, θα πούμε τη γνώμη μας και στο επόμενο θέμα. Υπάρχει λοιπόν μια αγωνία για να αναγνωριστεί η άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση ώστε να εξασφαλιστεί η ιδιωτική αγορά παροχής πιστοποίησεων. Πολύ φοβάμαι ότι το ζητούμενο αυτής της ε, προσπάθειας αλλά και το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας από αποστηρωμένα τεμάχια γνώσεων, έτοιμα για συναρμολόγηση, ανάλογα με τις εκάστοτε επιταγές της αγοράς και των κυρίαρχων οικονομικών συμφερόντων. Ο πληστηριασμός δεξιοτήτων θα λειτουργήσει ως μέσο πίεση των αμοιβών προς τα κάτω και θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας. Θα έχουμε δηλαδή υψηλές δεξιότητες με χαμηλές αμοιβέ. Η αξία λοιπόν της ολιστικής μάθησης και της ποιοτική δημόσιας εκπαίδευσης υποβαθμίζεται και τη θέση της παίρνουν οι ανάγκες της αγοράς, οι οποίες μέσω της συλλογής στατιστικών δεδομένων από την πλατφόρμα θα νομιμοποιούνται τελικά και θα καθορίζουν, θα κατευθύνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό με βάση την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η αναβάθμιση λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την άποψή μας του Europass που προτείνεται από την Κομισιόν υπερβαίνει κατά τη γνώμη μου το ίδιο το Europass. Ε, με την επιφύλαξη να καταθέσω συγκεκριμένες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα έρθουμε στους ε, πράσινους. Η Jill Lambert ε, από την Επιτροπή Απασχόλησης έχει το λόγο. Α, όχι, δεν είναι εδώ η Jill Evans τότε. Από τους πρασίνους. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους συγητές για το έργο που έκαναν για αυτή την έκθεση. Η πρόταση από την Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη βεβαίως και αντανακλά ακριβώς την επιτυχία του Europass και θα συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε μια, ένα καλύτερο και πιο προσβάσιμο και πιο σύγχρονο Europass για το μέλλον λόγω της αλλαγής των προποθέσεων στην αγορά εργασίας, των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε ε, το, να προωθήσουμε την αναγνώριση των δεξιοτήτων ε, και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούν πιστοποίηση των δικοτήτων που χρησιμοποιούν και οργανώσεις νέων για παράδειγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το, τις εισφορές το input όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Αλλά μοιράζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων σχέση με την ΕΣΚΟ. Είναι κάπως ε, πρόημο να χρησιμοποιηθεί η ΕΣΚΟ με τον τρόπο αυτό. Ε, χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω και να το εξάσουμε σε ένα μελλοντικό ε, σε μια μελλοντική στιγμή, αλλά όχι στην παρούσα φάση. Τώρα, όσον αφορά τις γλώσσες υπάρχει πρόταση να στις επίσημες ε, γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι βασικές επίσημες γλώσσες, γιατί όταν μιλάμε για προσβασιμότητα ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερες γλώσσες είναι δυνατό. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόταση είναι καλή, επιδέχεται βεβαίως βελτιώσεων, αλλά φαίνεται υπάρχει πλατιά συνένεση στην Επιτροπή και εγώ θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες ε, κάτω από αυτό το πρίσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η FTT δεν είναι παρούσα. Θα έρθουμε στην κυρία Πίλε. Εμένα με καθησυγάζει η δουλειά των δύο συνεισηγητών. Ε, το σχέδιο έκθεση για το Europass είναι πολύ λιγότερο ριζοσπαστικό από την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέτε καθαρά ότι το Europass δεν πρέπει να είναι μία ενιαία θηρίδα εκπαίδευση και κατάρτιση ε, και χαίρομαι για τη διευκρίνηση αυτή όσον αφορά τώρα το ΕΣΚΟ. Υποστηρίζω την προσοχή των εισηγητών. Η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι πολλοί επαγγελματίες ε, και ειδικότερα οι τοπικοί τεχνίτες και παραδοσιακοί τεχνίτες δεν μπορούν να ε, έχουν μια, έναν κοινό ορισμό. Ε, η εναρμόνιση των δεξιοτήτων δεν γίνεται να, είναι, να γίνεται με κίνδυνο την πολιτιστική ιδιαιτερότητα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να, χαρακ... να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας του Europass. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή θέλει να το καταστήσει ένα υποχρεωτικό εργαλείο, το οποίο όμως θα δημιουργήσει προβλήματα αναλογικότητας και επικουρικότητας. Παρά τις προσπάθειες που πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, η ομάδα μου δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή χωρών υποένταξη ή ενδεχόμενων υποψηφίων, οπότε από κοινού συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόληση για αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Τα συγκεκριμένα σημεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε σε άλλες παρεμβάσεις. Η συνάδελφος κυρία Σόντροβα από την ε, Επιτροπή Πολιτισμού. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο έκθεσης είναι ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο Το Ευρωπαϊκό Μέσο Κινητικότητας είναι νομίζω πολύ καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση, ε, αλλά νομίζω ότι μπορεί σαφέστατα να βελτιωθεί. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε την πρόταση των ε, εισηγητών ε, όταν λένε ότι πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό ε, που ε, θα κάνει το Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να αναβάλουμε την ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Γιατί ναι, μπορούμε να βιαστούμε, να αποφασίσουμε, αλλά θα ήταν πολύ πιο συνετό να περιμένουμε, να, να δούμε τι είναι αυτό που τελικά θα κληθούμε να τροποποιήσουμε. Είναι δύσκολο να τροποποιήσουμε κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Κύριε Μαν, λοιπόν, συμφωνώ απολύτως αυτό που είπατε να παραταθεί δηλαδή η ε, προθεσμία τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Για τα διαδικαστικά θα σας κάνω στο τέλος μία πρόταση. Η Julie Watch θα, πάρει, θα πάρει το λόγο και εάν δεν υπάρχει άλλο θα κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα Απλώς να πω κάτι καλό για το Europass, γιατί πριν πω στον πολιτικό στίβο εργάστηκα με νέους ανθρώπους οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι και δεν είχαν πρόσβαση σε πολλά από τα πράγματα που ίσως ε, άνθρωποι σε πιο προνομικές θέσεις έχουν. Και ε, ε, ορισμένοι υπάλληλοι στο επίπεδο των κοινοτήτων χρησιμοποίησαν το με του νέου ανθρώπου και θεωρούν ότι είναι χρήσιμο. Γι' αυτό εγώ συνεχίζω να ενθαρρύνω τη χρήση του Europass. Από μια προσωπική και πρακτική εμπειρία ε, το Europass είναι καλό εργαλείο, απλώς ε, χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω στην Επιτροπή τη δυνατότητα να μιλήσει. Κυρία Περεζίνη, είστε εδώ. Thank you, Chair. Η Επιτροπή καλωσορίζει τη σύνταξη αυτή της έκθεσης και ευχαριστεί τους συζητητές για αυτή την εργασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την, τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση και ενημέρωση του Europass όπως πρότεινε και η Κομισιόν. Λαμβάνουμε υπόψη τις τροπολογίες και τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα, ιδιαίτερα ως προς το, την ΕΣΚΟ και τις ανησυχίες των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Άρα ε, αναδιατυπώνεται το κείμενο από την Προεδρία δεν ήταν στην, στις προθέσεις μας να κάνουμε δεσμευτικό το Europass, όπως ισχύει για το ΕΣΚΟ. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε θέλουμε να εναρμονίσουμε τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεχόμαστε και τηρούμε την επικουρικότητα και αναγνωρίζουμε και την εργασία σε εθνικό επίπεδο. Εμείς προτείνουμε ένα μέσο το οποίο να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στη σημερινή πραγματικότητα που θα είναι χρήσιμο για τους τελικούς χρήστες. Ελπίζουμε λοιπόν το κείμενο να είναι σαφές, απλό και απλό και να έχει μια συγκεκριμένη στοχοθέτηση στους τελικούς χρήστες για να τους βοηθήσει. Για να το χρησιμοποιήσουν και να αντλήσουν ε, πλέον εκτήματα από αυτό. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να ε, προωθήσουμε, να προβάλλουμε γραφειοκρατία και διοικητικό και δημοσιονομικό φόρτο στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Περιζίνη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτή την πολύ γόνιμη συζήτηση για τις σχέσεις και τις δυνατότητες για περαιτέρω τροπολογίες. Θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω τους δύο συγητές αν θέλουν πάλι να πάρουν το λόγο, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να κάνω μία πρόταση και θα ήθελα να μου πείτε άμεσα τη γνώμη σας. Όταν το Συμβούλιο λέει ότι θέλει μια νέα πρόταση μέχρι τις 6, να την παρουσιάσει μέχρι τις 6 Απριλίου, είναι προφανές ότι δεν μπορούμε εμείς να κηρυθούμε σε μια άλλη κατεύθυνση, γιατί αυτό θα μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Είναι λοιπόν εύλογο εάν βάλουμε την 10η Απριλίου ως ημερομηνία, αλλά η πρότασή μας είναι να μην γίνει η εξέταση των τροπολογιών, για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την ε, προθεσμία στις 21 και 22 Απριλίου. Όχι, λέει η πρόεδρος, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει το Μάιο μάλλον, θα πρέπει να είναι Μάιος. Ε, η ημερομηνία για την ψηφοφορία, για να την ε, τηρήσουμε. Ε, ήταν λάθος αυτά που είχα στα χαρτιά μου. Ιούνιο η ψηφοφορία, προθεσμία 10 Απριλίου, 3 το μεσημέρι. Consideration of amendments, η εξάρτηση των δεν θα γίνει. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αρκετός χρόνος οι σκιώδεις να επεξεργαστούν κάποιες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες για το Europass, ίσως προς την ίδια κατεύθυνση που κινείται και το Συμβούλιο. Ο κύριος Μαν καταρχήν και μετά ο κύριος Μαλίνοφ. Καταρχήν ε, ευχαριστώ πολύ για την ευχάριστη είδηση ότι πραγματικά μπορούμε να ε, πάμε ως τη 10 Απριλίου. Νομίζω ότι είναι επικοδηματικό, είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή βάση. Ευχαριστώ πολύ και για τις ε, συνεισφορές στη συζήτηση. Η ΕΣΚΟ βρίσκεται σε πιλωτική φάση, δεν αξίζει να χρησιμοποιηθεί για το Europass. Ε, ε, και όσον αφορά το θέμα της μη υποχρεωτικότητας, μη θεσμευτικότητας. Και αυτό είναι σημαντικό. Ε, ε, όσον αφορά τους ορισμούς των δεξιοτήτων. Εδώ υπήρχαν ε, διαφορετικές ε, ε, προτάσεις. Θεωρώ ότι είναι καλό να πούμε ότι θέλουμε μία ενιαία αναθεώρηση και επιθυμούμε το Europass να εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό εργαλείο, εργαλείο σαν μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή η Ευρώπη έχει να προσφέρει ακόμα κάποια πράγματα και αν παραμείνει ο θελούσιος χαρακτήρας νομίζω ότι θέλουμε, έχουμε τη βάση την οποία επιθυμούμε. Ελπίζουμε λοιπόν στις 21 και 22 Ιουνίου να έχουμε κάτι το οποίο να μπορούμε να ψηφίσουμε με τη συνέντησή μας ήσυχη. Ο κύριος Μαλίνοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γενική η στάση μας ως ε, συγγητών ήταν αυτή που σας περιγράψαμε. Εγώ πάντως συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη ε, από τα σχέδια των κρατών μελών και να μας δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Αν όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ίσως θα έπρεπε λίγο να την εξομαλύνουμε και να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε και πιο ριζοσπαστικές προτάσεις όταν θα είμαστε έτοιμοι να τις εφαρμόσουμε. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να συγχαρώ τους ανθρώπους που είναι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια για την γενική τους ε, αίσθηση ότι το Europass όντως χρειάζεται αναθεώρηση, ειδικότερα ως προς τη συμπερίληψη κάποιων ε, μη ε, τυπικών προσόντων, κάποιων προσόντων εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ε, θεωρώ ότι το μέλλον θα βασιστεί πολύ σε τέτοιου είδους ε, εργασία και αν θυμάμαι, καλά, αυτό που θυμάμαι από αυτή τη συζήτηση είναι ότι ο όρος κοντά στην τελειότητα ε, χρησιμοποιήθηκε. Ε, βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να το πλησιάσουμε με την προσπάθεια που κάναμε για συμβιβασμό. αν είχαμε δεχθεί καθαρά τις προτάσεις των κρατών μελών δεν θα τα είχαμε καταφέρει και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παραγνωρίζει ότι τα, η διατύπωση και μόνο φόβησε πολλούς, ε, πολλούς φορείς στα κρατημέλη και αυτό δείχνει την ε, κατεύθυνση προς την οποία θα έπρεπε να κινηθούμε στο μέλλον. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν κάτι είναι υπερφιλόδοξο ή υπερβολικά ρηψοκίνδυνο, ε, καλό είναι να μας δίνεται και περισσότερος χρόνος να το σκεφτούμε. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι στο μέλλον που θα ασχοληθούν ακριβώς με αυτό το θέμα και το ΕΣΚΟ θα αποτελεί τμήμα του Europass και για να το υπερασπιστώ και όλα σε αυτό το σύστημα ήταν ένα σύστημα επιτυχημένο σε πολλές χώρες και μπορώ να αφαιρθώ τουλάχιστον την Ισπανία και τη Βουλγαρία όπου πραγματικά θεωρείται επιτυχημένο ε, με βάση σχεδόν οποιοδήποτε κριτήριο, όχι μόνο τον αριθμό των βιογραφικών, αλλά έχει αλλάξει την οτροπία των νέων, των εργοδοτών. Μπορώ να ε, δεν μπορώ να σας δείξω ούτε ένα ε, βιογραφικό τα τελευταία χρόνια που να μην είναι βιογραφικό Europass. Είναι τεράστια αυτή η αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις περαιτέρω εργασίες σας για ένα καλό μέλλον του Europass, καλές συζητήσεις με τους Κιώδης και μετά από τη σημερινή συζήτηση έχω την ελπίδα ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ και επαναλαμβάνω. Ε, συμφωνήσαμε 10 Απριλίου Τρεις το μεσημέρι η ημερμηνία κατάθεση τροπολογιών, η εξέταση τροπολογιών δεν θα γίνει και η ψηφοφορία είναι στις 21 και 22 Ιουνίου. Θαυμάσια λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα έρθουμε στο δεύτερο θέμα της κοινή μας συνεδρίασης για τη νέα skills agenda για την Ευρώπη. Οι συγητές είναι συνάδελφοι Λάμποβα και ο συνάδελφος Μόμσιλ, Νέκοφ, συγγνώμη. Και θα παρακαλέσω, θα δώσω το λόγο στη συνάδελφα από την Επιτροπή Επασχόλησης για τα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε στην ευρωπαϊκή μας ατζέντα. Είναι ένα κοινό θέμα των επιτροπών μας και χαίρομαι γιατί μπορέσαμε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Περνάει ο χρόνος, δεν έχουμε περιθώρια, γι' αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό το θέμα αυτό και να φτάσει στον τελικό χρήστη. Ε, δίνω το λόγο στην κυρία Κλαβαγιώβα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου αναθέσατε αυτή την έκθεση. Ε, είμαι κοινή συντάκτρια μαζί με τον κύριο Νέκοφ. Μιλάμε για νέες δεξιότητες και χαίρομαι που δουλεύω με έναν νέο ευρωβουλευτή, πολύ νέο, γιατί έχει άλλη ε, θεώρηση του ζητήματος. Ε, χαίρομαι που οι δύο μας επιτροπές συνεργάζονται και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεδριάζουμε από κοινού. Γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχει απασχόληση χωρίς εκπαίδευση και τούμπαλιν. Η συνεργασία μας με τον ε, συνεισηγητή ήταν πολύ καλή. Είδαμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητας. Βεβαίως η έκθεση δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί υπάρχει δυσκολία ως προς τον ε, χώρο και το χρόνο. Εγώ από πλευράς ε, Επιτροπής Απασχόλησης θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία και να σας πω την άποψη της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για θέσεις εργασίας σημαίνει ότι οι δεξιότητες που δίνουμε στους ανθρώπους σχετίζονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Δηλαδή η μάθηση θα πρέπει να σχετίζεται με τις ανάγκες της ε, αγοράς. Θα πρέπει να είναι δεσμευτική δεσμευτικό τμήμα της εκπαίδευσης και να υπάρχει και μία πρώτη, πρώτη επαφή με τους ενδυνάμει εργοδότες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, λάβουν υπόψη την επιχειρηματική εκπαίδευση στο πρόγραμμα διδακτέας ε, ύλης και να προωθήσουν και την αρχή δεξιοτήτων. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης. Θεωρώ ότι η κοινωνική εταίρη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα για να ορίσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και δεξιότητες που σχετίζονται με αυτές τις ανάγκες. Άρα θα πρέπει να προτρέξουμε ως προς τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς για να προσδώσουμε στους μαθητευόμενους και τη δυνατότητα για να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες. Χρειάζεται ένας μηχανισμός ίσως δεξιοτήτων για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, βλέπουμε από τις βέλτιστες ε, πρακτικές των κρατών μελών ότι οι χώρες που έχουν καλά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν ε, χαμη... χαμηλότερο, χαμηλότερο δίκτυο ανεργίας. Άρα θα πρέπει να διδαχθούμε από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, γιατί πολλές φορές μιλάμε για αυτές τις πρακτικές, αλλά δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να ε, ε, λάβουμε υπόψη τις δεξιότητες αυτές, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για να γίνει η αγορά πιο δελεαστική για τους ανθρώπους. Ε, δέχομαι την ατζέντα δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω η Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δικές μας συστάσεις και εύχομαι να συνεργαστώ με όλους σας ε, για αυτή τη σημαντική έκθεση γιατί σκεφτόμαστε για το τι μπορούμε να κάνουμε για τις μελλοντικέ γενναίες. Σας ευχαριστώ πολύ και με μεγάλη χαρά θα συζητήσω περαιτέρω ζητήματα με τον συνεισηγητή. Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Nekov. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λέκοφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ουλσκογ. Θα ήθελα να πω και εγώ ορισμένα πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σλαμπάγεβα πραγματικά. Είναι μια μεγάλη χαρά να δουλεύουμε μαζί της και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα στο μέλλον. Η δουλειά μας ήταν πολύ οργανωμένη και νομίζω ότι η έκθεσή μας είναι πολύ υψηλή ποιότητας. Περιμέναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα για αυτό το νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες. Και τώρα αυτό το θεματολόγιο θέτει πάρα πολύ σωστά το θέμα, λέγοντας ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέες δεξιότητες, γιατί το περιβάλλον εργασίας μας και η αγορά εργασίας μας αλλάζει. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά εστιάζει στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Εμείς πιστεύουμε ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα πρέπει να μπορούν να προσπαθούν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες για τους νέους, να τους διδάσκουν την κριτική σκέψη, το κριτικό πνεύμα και τη λήψη αποφάσεων με, με κριτικό πνεύμα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει πολλά προβλήματα. Προτείνονται και νέες στρατηγικές όσον αφορά την εργασία με χαμηλές, ε, χαμηλό επίπεδο δεξιότητες. Το 2025, 40% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτούν υψηλού επίπεδου δεξιότητες, 40% ε, μεσαίου επίπεδου και μόνο 11% χαμηλού επίπεδου. 40% των, εργαζομε... των εργοδοτών συγγνώμη, θεωρούν ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία δεξιοτήτων ε, στην αγορά εργασίας. Από την άλλη, οι χαμηλού επίπεδου δεξιότητες, ε, ε, χαμηλού επίπεδου εξωτείων εργαζόμενοι έχουν δυσκολία να βρουν εργασία. Όσον αφορά τις λεγόμενες ανάγκες των νέων, η ανεργία είναι στα ύψη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ περίπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν ε, ανάγνωση και μαθηματικά και συνεπώς δεν έχουν ε, ένα αξιοπρεπές ε, βιωτικό επίπεδο. Η ψηφιοποίηση είναι ένα ακόμη ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσω. Αλλάζουν τα πάντα με την ψηφιοποίηση. Αλλάζει ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που διδάσκουμε και μαζί με την κυρία Σλομπάγεβα εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια πιο οριζόντια προσέγγιση βάσει της οποίας ε, οι σπουδαστές ε, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Υπάρχει κάτι που απουσιάζει από την ανακοίνωση, δεν εστιάζει επαρκώς ε, στους, σε όσους εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς ε, και στην προσχολική ηλικία και τη σχολική ηλικία. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα ώστε να επιτύχουν τους στόχους της Βαρκελόνης. Το 30% των παιδιών κάτω των τριών πρέπει να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα το, το, το νωρίτερο δυνατόν. Η εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό λοιπόν το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων πιστεύω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην διαβίου μάθηση. Ξέρουμε ότι σήμερα οι εργοδότες ε, ζητούν και ήπιες δεξιότητες. Μόνο 25% των, των εργοδοτών ε, προσφέρουν ε, περιόδους μαθητείας. Θα ήθελα να πω και ορισμένα πράγματα σε σχέση με την επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση. Σε μερικές χώρες ε, εξελίσσεται πολύ καλά ε, αυτό κατόπιν συστάσεων που έγιναν πριν από μερικά χρόνια. Και υπ' αυτήν την έννοια νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο μεγαλύτερη πολιτική βούληση. Αυτή η επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις χώρες γιατί επιτρέπει στις ε, χαμηλού επίπεδου δεξιοτήτων ε, ε, ε να συμμετέχουν και ο στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Η κυρία Σλοπάγεβα είπε ότι ότι η δυτή εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να εργάζεται ενώ σπουδάζει. Και με αυτή την ευκαιρία μαθαίνουν πολύ περισσότερο για αυτά που απαιτούνται στην αγορά εργασία. Και θα ήθελα τέλο να πω ότι πρέπει να επενδύσουμε όχι μόνο στην ψηφιοποίηση και στην υποδομή, αλλά και στους διδάσκοντες. Πρέπει και εκείνοι να διδαχθούν πώς θα χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία. Και ο στόχος δεν είναι μόνο οι βασικές δεξιότητες για τους σπουδαστές στην Ευρώπη. Θέλουμε να κατέχουν καλύτερα τα βασικά ε, ε, τις, βασικές ε, τα, βασικά μαθήματα και χρειαζόμαστε και διαβίου μάθηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο εισηγητές και τώρα θα περάσουμε στους ε, σκιόδους για δύο το πολύ τρία λεπτά και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Σόντροβα η οποία θα μιλήσει εξ ονόματος τόσο του πολιτισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού όσο και της ε, ε, Πασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για μια έκθεση η οποία επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο είναι σημαντικό, δηλαδή απασχόληση και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι ε, ε, ενισχύουν αυτό το οποίο προτείνει η Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα. Υποστήριξη του διτού εκπαιδευτικού συστήματος, επαγγελματική κατάρτιση και συνεργασία με τη συνεργοδοσία η συνεργασία με την εργοδοσία είναι σημαντική όχι μόνο στην προπαρασκευαστική φάση, αλλά επίσης όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια μεταγενέστερη φάση. Επίσης ε, υπογραμμίσατε την πρώιμη μάθηση, την προσχολική μάθηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παραγνωρίσει η Επιτροπή και νομίζω ότι είναι θετικό ότι το επισημαίνεται. Επισημαίνεται επίσης τη σημασία της επίσημης και ανεπίσημης ε, εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό ότι το διαχωρίζεται σε ένα χωριστό κεφάλαιο και ο κύριος Νέκοφ αναφέρεται στον ε, στόχο ενός ε, διατύπωσης νομοθετικού πλαισίου σε κάθε χώρα. Στη Τσεχία έχουμε ένα νόμο για την αναγνώριση ε, της, ε, το αποτελέσμα της επαγγελματική κατάρτισης. Ε, όπως είπατε, ε, η εργοδοσία, της άτυπης ε, κατάρτισης. Όπως ε, είπατε, η εργοδοσία έχει κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την αναγνώριση της ανεπίσημης εκπαίδευσης. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το επιβάλλουμε στις χώρες μέλη, απλώς να το προτείνουμε σαν εργαλείο. Την άτυπη εκπαίδευση θα μπορούσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε αυτό το νόμο λοιπόν στην Τσεχία και θα μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε τις θετικές και τις αρνητικές μας εμπειρίες εδώ. Πρόκειται Όσον αφορά τους διδάσκοντες και εδώ δεν εξετάζεται επαρκώ ο ρόλο τους. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες όπως προτείνει η Επιτροπή θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, εκπαίδευση και υποστήριξη των διδασκόντων. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια πιο ειδική πρόταση εδώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πει προς τις χώρες μέλη ότι θα πρέπει να, τους υποστηρίξει όσον αφορά την υποστήριξη των διδασκόντων, γιατί η επαγγελματική κατάρτιση για την επαγγελματική κατάρτιση οι διδάσκοντε δεν είναι παρκώ προετοιμασμένοι. Όσον αφορά τη διαβίου μάθηση, την εκπαίδευση των ενηλίκων, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Πρόκειται για ένα τρόπο ε, διαδίδοντας την, ε, να διδώσουμε την ιδέα ότι αναγνωρίζουμε την αξία της εκπαίδευσης αυτή καθ' αυτή. Και χθες ε, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή για τα αποτελέσματα της μελέτης PISA. Στην Ευρώπη υπάρχουν 20% των μαθητών, ένα κομμάτι, το 20% των μαθητών ε, δεν έχουν τις βασικές ε, δεξιότητες. Εμείς δεν θέλουμε μαθητές ε, να καταλήξουν άνεργοι και στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν εργαλεία ούτε ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ήμουνα πιο γενναιόδορη στην κυρία Σόντροβα γιατί μίλησε εκ μέρους δύο επιτροπών. Οι άλλοι θα πρέπει να τηρήσουν το περιθώριο των δύο λεπτών. Ο κύριος Πάβελ έχει το λόγο από την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρτίνα Ντελαμπάιωβα και τον κύριο Νέκοφ για την εργασία τους Πολλά προελέχθησαν στις δηλώσεις σας, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή η ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη είναι κάτι το καινοτόμο και θα πρέπει να δούμε τι εργασία γίνεται στα κράτη-μέλη και ανά την Ευρώπη για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δεξιότητες που ορίζονται με βάση τις ανάγκες των πολιτών εκτός και εντός αγοράς εργασίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την πλήρη δέσμευση των κρατών μελών. Αυτό είναι εκ των νόνουκ άνευ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νέες ε, τεχνολογικές δεξιότητες του 21ου αιώνα ή και τις βασικές δεξιότητες όπως ανέφερε ο Μουντσι Νέκοβ, έτσι ώστε το σύστημα εκπαίδευσης να μπει σε μία φάση νέας ε, νιώτης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το πλαίσιο διαπραγματεύσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή με συγκεκριμένα μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann... Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε στην άνθρωπο κυρία Σιτένσκα από την Επιτροπή Απασχόλησης και το ECR. Sprechen auch wieder mit für Herrn Lohr. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για μια πραγματικά πολύ καλή έκθεση. Επετέλεσαν πολύ καλό έργο και συμφωνώ σχεδόν με όλα. Είναι σημαντικό στον κόσμο αυτό να προσανατολιστούμε προς τις νέες ε, δεξιότητες, τη διαβίου μάθηση, και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι αναγκαίο επίσης να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και εκτός δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί αυτό οδηγεί σε μια καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Επίσης είναι σημαντικό να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας ανθρώπους που είναι υπερχρεωμένοι και οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια δυσκολία και όταν εργάζονται δεν τους ε, μένει απολύτως ε, τίποτα στην τσέπη. Τώρα, για να μιλήσουμε περαιτέρω για δεξιότητες, δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε κάποιες ε, φάσεις που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω εξέλιξη στα σχολεία και στην ε, ζωή με τα παιδιά με αναπηρίες κυρίως. Είναι σημαντικό να ε, συγκεντρωθούμε εδώ στην καλύτερη κατάρτιση των ε, διδασκόντων ούτως ώστε να μπορούν να εργάζονται με παιδιά που έχουν ειδικέ ανάγκες ή εμφανίζουν αναπηρίες. Τέλος, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, να ρίσω μάλλον κάτι το οποίο αναφέρεται στην έκθεση. Το ζητούμενο είναι η διαβίω μάθηση όχι μόνο για τους ανέργους αλλά και για τους εργαζόμενους. Είναι σημαντικό όλοι να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύονται στο διηνεκές ούτε ώστε να μην να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα. Γιατί η υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερες ε, δυσκολίες ε, να ε, επιμορφωθούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιες μορφές άτυπης εκπαίδευσης που να υποστηριχθούν και από τους εργοδότες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ηγητές για το έργο τους θεωρώ ότι ε, εμείς στο ECR ε, έχουμε μια ολιστική προσέγγιση βασισμένη στις βέλτιστες ε, πρακτικές. Δεν είμαστε υπέρ υποχρεωτικών μέτρων γιατί το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες των χωρών μελών. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντας στο προηγούμενο θέμα, κάποια στιγμή έβαλα έναν αστερίσκο και είπα για την πολιτική δεξιοτήτων, θα μιλήσω στο δεύτερο θέμα, δηλαδή τώρα. Η συζήτηση λοιπόν για το νέο θεματολόγιο των δεξιοτήτων μου δίνει την ευκαιρία να πω τις σκέψεις μας και για την έκθεση. Ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές. Επιτρέψτε μου λίγο και τον προσωπικό τόνο. Ε, ε υπογραμμίζω ότι οι συγητές μας είναι και δύο νέοι άνθρωποι και επομένως τα θέματα εκτός από την πολιτική κομματική θέση τα ζουν βιωματικά τα προβλήματα των νέων αυτά που, και ιδιαίτερα το πρόβλημα της απασχόλησης, της ανεργίας, της ανάπτυξης επομένως τις παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις οποίες διατυπώθηκαν. Πριν με ευχαριστήσουν, ακούστε τις παρατηρήσεις μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα, αυτό το θέμα αφορά πράγματι και το παρόν και το μέλλον. Αφορά τις νέες γενιές. Ε, Πράγματι η τεχνολογική πρόοδος, η ανάπτυξη, η επικοινωνιακή πολιτική, τα νέα δεδομένα, έχω σπουδάσει θετικέ επιστήμες και κοινωνικέ επιστήμες, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να τα πάρουμε υπόψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η συζήτηση όμω αυτή για τι δεξιότητε και για την κατάρτιση με αφορμή το θεματολόγιο δεν μπορεί να ξεκοπεί από την, τη συζήτηση τι Ευρώπη θέλουμε. Δηλαδή τι είδου κοινωνίες θέλουμε και τι είδο μοντέλο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον επιθυμούμε μέσω αυτών των παρεμβάσεων. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά και σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο έκθεση που σχολιάζουμε δεν αμφισβητεί το οικονομικό μοντέλο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να ενισχύσει μέσω του συγκεκριμένου θεματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, δεν αφισβητείται η Ευρώπη των δύο και τριών ταχυτήτων που έχει δημιουργηθεί. Δεν αφισβητούνται οι πολιτικέ γενικευμένη λιτότητα που εφαρμόζονται σε πολλά κράτη. Δεν αφισβητούνται οι πολιτικέ που προωθούν την απόκληση αντί τη Και εδώ επιτρέψτε μια επίκαιρη αναφορά. Εκτός αν για τα προβλήματα, τα προβλήματα της ενεργείας, τα οικονομικά που παρουσιάζονται κυρίως στις χώρες του Νότου, ισχύει η ερμηνεία του κύριου Ντάζευλου. Και επειδή είμαστε επιτροπές πολιτισμού και παιδείας, να πω ότι οι Ευρωπαίοι χωρίζονται στους οπαδούς του Φιλίδωνου αρχαίου Θεού Διονύσου ή οπαδούς του Καλβίνου. Δεν ξέρω αν αυτά θα υποθούν στην εκπαίδευση, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είναι αυτή η αιτία, έχει, όμως η αιτία είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές τις οποίες υλοποιεί και αυτή η πολιτική των δεξιοτήτων, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πάμε στο σωστό μοντέλο. Έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που προωθεί μεγάλες αποκλήσεις στην οικονομική και τη βιομηχανική ανάπτυξη, στα επίπεδα και τα ίδια ανεργίας και το προτινόμενο θεματολόγιο όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά κατά την άποψή μου βεβαίω θα, οξύνει, θα το οξύνει λειτουργώντας ως διάβλος μετακίνησης, διοχέτευσης εργατικού δυναμικού από ορισμένα κράτη-μέλη σε άλλα, πράγμα που το βλέπουμε και γίνεται εκ των πραγμάτων με το brain drain που έχουμε σχολιάσει αρκετέ φορέ. Στα κείμενα, ε, κατά την άποψή μου, προωθείται η εργασιακή ανασφάλεια, ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο και καθορισμένο τη τι επιταγέ τη αγορά, η χρήση αορίστων ενιών, όπω η επιχειρηματικότητα και κινητικότητα και ω πανάκια για το πρόβλημα τη ανεργία των νέων. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν τίθεται τα ζητήματα των εργασιακών δικαιωμάτων και δεν άκουσα από την Επιτροπή Απασχόληση του Κοινοβουλίου τι γίνεται με τι συλλογικέ συμβάσει, τι γίνεται με τα εργασιακά δικαιώματα. Πανάκια είναι η επιχειρηματικότητα, μια όριστη έννοια ή η κατοχήρωση ορισμένων ε, δικαιωμάτων που με αγώνε έκαναν. Και πρέπει να τα εξασφαλίσουμε και στου νέου ανθρώπου, λέγοντα ότι με τι νέε δεξιότητε, απορριθμίζοντα την αγορά εργασία, απελευθερώνοντα τι αγορέ αυτό είναι η προτεραιότητα και στην εκπαίδευση. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το λύσει το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Σταματώ εδώ. Κυρία Πρόεδρε, τα είπα αυτά που ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στους πρασίνους. Κυρία Λάμπερτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συνεισηγητές για τη δουλειά τους. Τι θα θέλαμε να προσθέσουμε. Κάτι που, είπε, κάτι που γράφει και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρεται όχι μόνο στην μελλοντική αγορά εργασίας και την μεταρρύθμιση της που καλύπτεται πολύ καλά στην έκθεση, αλλά και τη μετάβαση σε μια κυκλική και χαμηλής περιεκτικότητα σε άνθρακα οικονομία που σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζεται η αγορά εργασίας στα προφίλ ε, των θέσεων εργασίας που ε, είναι αναγκαία. Νομίζω ότι μπορούμε να το ενισχύσουμε στην έκθεση γιατί αναφέρεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί όσον αφορά τις ε, δεξιότητες πολύ καλά αναφέρονται, αλλά δεν υπάρχει επαρκές πλαίσιο βιωσιμότητας που να αναφέρεται, που είναι κάτι που θα είναι σημαντικό για το μέλλον. Όσον αφορά αυτά τα STEM skills, τις ε, κύριες δεξιότητες, ε, καταλαβαίνω βέβαια ότι πρέπει να τηρήσουμε και τον περιορισμό χαρακτήρων ε, στη Κοινοβούλιο, αλλά αυτό το θέμα των STEM skills των βασικών κυρίων δεξιετήτων, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε περισσότερο. Επίσης μπορούμε να ενισχύσουμε και το ε, κομμάτι εκείνο που αφορά την ευθύνη των εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων και άλλων παρόχων, να υπάρχει κινητικότητα εντός των τομέων, που θεωρώ ότι είναι τμήμα ε, της ε, ε, πρόθεσης στην προσπάθεια αυτή και τα σημεία επανεισόδου στην αγορά εργασίας, το οποίο το είπε και συνάδελφος από την ECR, μερικές φορές χρειάζεται ο κόσμος να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας, σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης και πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Το ερώτημα επίσης που αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, την ποιότητα των ε, σχέσεων, των, ε, της μαθητείας. Ε, το Ίδρυμα Δουβλίνου έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά για αυτό το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση γιατί θεωρούν ότι δεν τους καλύπτει σε σχέση με αυτά που θα χρειαστούν για το μέλλον τους. Πώς είναι δυνατόν να δούμε την πιο δημιουργική διάσταση των δεξιοτήτων που είναι κάτι που ε, εξαιρετικά σημαντικό για τη ε, ζωή των ανθρώπων όπως και για την εργασία τους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Evans από την Επιτροπή Πολιτισμού και τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια καλά σημεία στην έκθεση και συμφωνώ με την έμφαση που δίνεται στην ανάγκη να βελτιωθεί η επαγγελματική κατάρτιση και η άτυπη εκπαίδευση που είναι σημαντική για να καλυφθούν τα ελλείμματα δεξιοτήτων που έχουμε στην οικονομία μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη να αναπτύξουν ε, σωστά τις δεξιότητες ε, και να το δούμε αυτό, όποιες δεξιότητες και αν είναι αυτές. Επίσης, η ανάγκη ε, να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Οι δράσεις για το περιβάλλον θα πρέπει να συνδεθούν με την ανάπτυξη κάποιων συγκεκριμένων δεξιοτήτων και να συμπεριφθούν στο θεματολόγιο. Επίσης, η εκπαίδευση, ε, η κατάρτιση μάλλον, η εκπαίδευση των ενεργών πολιτών ε, σε σύνδεση με τις γλωσσικές δεξιότητες. Γλωσσικές δεξιότητες και όσον αφορά τις μειονοτικές ε, γλώσσες και κάλυψη των αναγκών των μεταναστών. Εγώ θα καταθέσω κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ και πάλι τους συγητές. Ε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Εύανς. Και ολοκληρώνοντας το γύρο των σκιωδών, η κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα σημεία. Θα θέλαμε να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους με αναπηρία και τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Πριν εντάξουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μιλάτε για διαφυγή εγκεφάλων, αλλά βλέπετε ότι υπερισχύει η λογική της αγοράς και όχι τα συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα κρίνουν τι είναι καλό ή τι δεν είναι καλό για αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθουμε τώρα στις λοιπές ναι. ε, παρεμβάσεις. Παρακαλώ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Η κυρία Γιαλοβλάκα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για μια πραγματικά άψογη έκθεση. Και θα ήθελα να πω τα εξής. Οι ψηφιακές δεξιότητες, μια ευέλικτη προσέγγιση είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εγώ είμαι υπέρ της διεύρυνσης του καταλόγου των δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε στρατηγική σκέψη, διαχείριση των γνώσεων, ομαδικό πνεύμα, ε, ε, δεξιότητα λήψη αποφάσεων, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ε, σαφήνεια της, την ενημέρωση, της, της πληροφορίας, την πληροφόρηση. Ε, όλα αυτά είναι στρατηγική σημασία. Οι διδάσκοντες ε, εκ παραδόσεω παραδίδουν γνώσει. αλλά σήμερα θα πρέπει οι διδάσκοντες να διδάξουν τους διδασκόμενους πώς μπορούν να επαληθεύουν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους γιατί πολλές φορές οι πληροφορίες, τα δεδομένα περιλαμβάνουν ε, ψεύτικα κατασκευασμένα νέα κηρύγματα μίσους κλπ. Οι νέοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο σεβασμό, στους τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους και πραγματικά Αυτές είναι δεξιότητες οι οποίες ε, βρίσκονται σε φθήνουσα πορεία και νομίζω ότι είναι σημαντικό στο σχολείο να μπουν στο επίκεντρο της εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, μιλήσω για την προοπτική της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίσουμε θέματα ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Άρα θα πρέπει να δούμε τις ψηφιακές δεξιότητες, όχι μόνο από την πλευρά των εργαζομένων, αλλά και των πελατών και των πολιτών. Εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή ως προς τις ε, ψηφιακές δεξιότητες, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας σε έναν ψηφιακό κόσμο. Τώρα νομοθετούμε για την ιδιωτικότητα και για την προστασία των δεδομένων. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνένεση των ε, πελατών. Αλλά οι πελάτες που δεν έχουν αυτή τη γνώση δεν μπορούν να προβούν και στη σωστή επιλογή. Και αυτή η οριοθέτηση δεν υπάρχει στις ψηφιακές δεξιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες να μπορούν να αποτιμηθούν από τους πελάτες και από τους καταναλωτές. Vielen herzlichen Dank. Ο κύριος Μαν, ευχαριστούμε πολύ τους νεαρούς ε, εισηγητές. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί πολλοί στη συνέχεια δεν έχουν καμία ευκαιρία. Ε, στη Γερμανία υπάρχει μια φρικτή, ένας φρικτός κοινωνιολογικός όρος παιδιά από οικογένειες ε, που είναι ε, απομακρυσμένες από τον ε, εκπαιδευτικό χώρο, αυτό σε μία έννοια, σε μία λέξη. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε ούτως ε, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ε, ολοκληρώσουν τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί δεν θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εγκαταλείπονται στην τύχη τους αν έχουν ε, εγκαταλείψει το σχολείο. Επειδή Αντιπρόεδρος θα φύγει, θα ήθελα να της δώσω συντομία το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Πέτρα, και όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας, ε, γιατί ε, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Έχουμε ένα κοινό θεματολόγιο και μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης που βρίσκονται εδώ ότι στις 10 και 45 θα συνεχίσει η δική μας συνεδρίαση την οποία διακόψαμε χτες το απόγευμα εθουσα 6 6Q2. Εγώ θα φύγω τώρα και θα πάω στην αίθουσα της συνεδρίας γιατί έχουμε πολλά σημαντικά θέματα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνεδρίαση. Και από τη δική μου πλευρά σας ευχαριστώ. Νομίζω θα συνεχίσουμε αυτή την πραγματικά καλή μας και δοκιμασμένη συνεργασία Ελπίζω τα μέλη της Επιτροπής της Απασχόλησης να βρουν τον δρόμο για την 4Q2. Η Julie Ward έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πέτρα. Συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να πω πόσο σημαντικό είναι οι δημιουργικές ε, δεξιότητες να συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε θεματολόγιο στη συνέχεια, γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και μέσω της δημιουργικότητας μπορούμε να ζήσουμε μαζί, μαθαίνουμε τη συνεργασία ε, και αποκτούμε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ε, το να μαθαίνει κανείς για την τέχνη δεν ε, είναι μόνο για την ίδια την τέχνη, αλλά για ολόκληρη τη ζωή. Νομίζω ότι και η διαβίου μάθηση μπορεί να συμπεριλάβει ε, την συνδικαλιστική ε, διαδικασία. Εμείς έχουμε τον ε, οργανισμό μάθησης των εργαζομένων ε, που ουσιαστικά μαθαίνει στους εργαζόμενους πώς να συνδικαλίζονται. Επίσης υπάρχει και το θέμα του επαγγελματισμού του επαγγελματικού αλφαβητισμού. Είναι μια νέα ιδέα που μπορεί να μας βοηθήσει στο να κινηθούμε προς τα εμπρός και είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των μεταναστών, των προσφύγων που δημιουργούν, που επιφέρουν νέες δεξιότητες, εμπλουτίζουν τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες μας. Η δική μας ε, η ε, η δική μου οι προ, ε, ήταν ε, Γάλλοι από τη Βόρεια Γαλλία οι οποίοι έφεραν πάρα πολλά καινούργια πράγματα στην Αγγλία και τελικά ε, συνεισέφεραν στον πλούτο της πόλης στην οποία κατέληξαν ερχόμενοι από την Νότια Γαλλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χτες κυρία Πρόεδρε κάποιοι στο Λονδίνο έχασαν τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο μιας τρομοκρατικής επίθεσης και κανένας δεν το είπε σήμερα ε, κάποιοι από τους τραυματίες ε, ε, είναι μαθητές, σπουδαστές που δεν είναι μόνο Βρετανοί, είναι Γάλλοι και Ρουμάνοι. Πρέπει πραγματικά να το λέμε και αυτό, για μένα είναι πολύ έντονο αυτό συναισθηματικά. Καθόμαστε εδώ και συζητάμε για τους νέους και δεν είπαμε τίποτα για τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν στο Λονδίνο και που τραυματίστηκαν. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο εν συντομία στην Επιτροπή. Ε, σύντομα παρακαλώ, γιατί οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να περπατήσουν πολύ ώστε να φτάσουν στην αίθουσα της συνεδρίας τους. Ευχαριστώ πολύ και ε, ευχαριστούμε για την ε, ε, έκθεση. Η Επιτροπή προσεγγίζει, χαιρετίζει την έκθεση και τις προσπάθειες των χωρών. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, εδώ γίνεται μνήα στην έκθεση, αλλά διερωτώμεθα κατά πόσο θα ήταν παρόλα αυτά δυνατόν να ταξινομηθούν κάπως οι δεξιότητες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, είναι σαφές ότι η skills agenda δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση και είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, προβλέπει επιπλέον ε, χρηματοδότηση και στο πλαίσιο του Erasmus ε, Plus και άλλων προγραμμάτων και θα ήταν σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ και επειδή ξέρω ότι θα πρέπει να φύγει, θα ξεκινήσουμε την κυρία Λαμπάγιοβα. Θα έχουμε και άλλες συνεδριάσεις μαζί, οπότε θα καταφέρετε να προφέρετε καλύτερα και το επώνυμό μου. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπατε συνάδελφοι. Επειδή αναφερθήκατε στις βέλτιστες πρακτικές, τα κίνητρα των κρατών μελών, τα μέσα που είναι στη διάθεση των κρατών μελών, ε, την ε, ε, κατάρτιση των διδασκόντων που είναι πολύ σημαντική, επιχειρηματικές δεξιότητες, οικονομικές δεξιότητες ως προς την προσέγγιση στη ζωή, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι δημιουργικές δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βόρτ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να υποβάλουμε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και το αποτέλεσμα αυτών θα φανεί σε 10 χρόνια. Ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα με την εκπαίδευση. Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα για να έχουμε τα αποτελέσματα σε 10 χρόνια. Αυτό, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να δράσουμε τώρα. Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, όλα, όλα τα καλά λόγια που είπατε. Ε, εγώ συνεργάζομαι με νέους συναδέλφους, γι' αυτό φαίνομαι νέα. Και νιώθω και καλύτερα. Σας το προτείνω, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα να το κάνετε κι εσείς. Έτσι θα νιώσετε κι εσείς νεότεροι δεν είναι, είμαστε μόνο νέοι, αλλά είμαστε και δημιουργικοί. Οπότε σκεφτόμαστε να οργανώσουμε μια ειδική εκδήλωση, μια ακρόαση, αν οι επιτροπές, οι πρόεδροι των επιτροπών και οι γραμματείες συμφωνήσουν, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να προσκαλέσουμε διδάσκοντες, εργοδότες, νέους, ε, που να μας παρουσιάσουν πολύ συγκεκριμένα κάποιες προτάσεις, για να ακούσουμε από, το, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους συγκεκριμένες προτάσεις. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα συμπεράσματα στην έκθεσή μα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα είμαστε και δημιουργικοί στη σκέψη μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ε, αναμένω συνεργασία με όλου σα. Ευχαριστώ πολύ και ο κύριος Νέκοφ παρακαλώ την συντομία. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα λάβουμε υπόψη μας ε, όλα τα σχόλια, όλες τις παρατηρήσεις με την κυρία Ντλαμπάγιοβα. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πραγματικά για την εξαιρετική μας ε, συνεργασία και τα σχόλια των συναδέλφων για την έκθεση. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Λάμπερτ όσον αφορά τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν βρίσκεται εδώ κυρία Λάμπερτς αλλά παρόλα αυτά θα πω ότι Χρειαζόμαστε υψηλά εδικευμένους ε, ανθρώπους προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν εντός αυτής της κυκλικής οικονομίας. Αυτό το οποίο συζητούμε εδώ ε, βεβαίως δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και θα ήταν μόνο ευχολόγιο εάν ε, δεν αποδεσμεύσει η Επιτροπή κάποια κονδύλια. Το Εράσμους και το και άλλα, ε, το έχει ήδη, τα κονδύλια του Εράσμος έχουν ήδη επιμεριστεί μεταξύ των χωρών μελών. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι η ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων και η ενίσχυση μιας, ε, ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης στην πλευρά των διδασκομένων και των διδασκόντων θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για μα. Θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον μα. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για όλα σας τα σχόλια και θα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά στο κείμενό μας και ε, πιστεύω ότι θα έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική έκθεση στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Όπως σας είπα, η πληροφορία θα γίνει τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης, καλές περαιτέρω διαβουλεύσεις και τα μέλη του, της Επιτροπής Πολιτισμού παρακαλούνται να παραμείνουν στην αίθουσα γιατί θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξή μας. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Καλημέρα σας.